Να το πείτε στον κύριο Σβόμποντα, κύριε Πόσελτ, που προεδρεύει στην ομάδα εργασίας. Ψηφίζουμε. Πάρτε τις κάρτες ψηφοφορίας σας, παρακαλώ. Έχω 7 προτάσεις για ψηφίσματα για το Πακιστάν. Θα ψηφίσουμε πρώτα για το Πακιστάν, για τη δολοφονία του κυβερνήτη του Πουντζάμπ, του κ. Τασίρ. Κοινή πρόταση ψηφίσματος, λοιπόν, παράγραφη 8 έχουμε προφορική τροπολογία που θα παρουσιάσει η κυρία Σάκε. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Η παράγραφος 8 θα πρέπει να προσθεθεί μετά το τέλος της παραγράφου 7 όπου θέλουμε να μπει η μνήμα να αποσύρουμε τους ενδιασμούς μας περί. Αυτό είναι η τελική μας πρόταση για το κείμενο. Αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Μπορούμε να το ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 4 έχουμε τα τμήματα ψηφοφορία και πάλι προφορική τροπολογία από τον κύριο Τάνοκ θα παρουσιαστεί. Ναι, ήθελα η παράγραφος 14 να αλλάξει ω έχει. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς την κυβέρνηση του Πακιστάν να προχωρήσει σε πλήρη αναθεώρηση του νόμου ε, κατά της βλασφημίας συμπεριλαμβανομένων και των ισοβίων καθήρξεων και την θανατική καταδίκη για οποιοδήποτε κριθεί ένοχος βλασφημίας κατά του προφήτου ε, ε, ε ακόμη και την ε, επανέναρξη της υπηρεσίας, ε, της λειτουργίας της υπηρεσίας για τις υποθέσεις ε, παραβιάσεων δικαιωμάτων μειονοτήτων. Ωραία. Αφού δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Υπέρ, για το πρώτο τμήμα, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε και ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 15. Και πάλι κατά τμήματα ψηφοφορία σε δύο τα Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 17. Άλλη μια προφορική τροπολογία. Κυρία Σάκε. Διάβασα και τα δύο. Άρα ισχύει αυτό που είπα στην προηγούμενη παρέμβασή μου, όπου ανέγνωσα και τα δύο τμήματα. That case we will... Πρόεδρος. Άρα θα ψηφίσουμε τώρα στο σύνολό του. Το ψηφίσμα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. So next item. Ακολουθεί, ακολουθούν μάλλον έξι προτάσεις ψηφισμάτων για την Βραζιλία και ειδικότερα για την έκδοση του Τσέζαρη Μπατίστη. Έχουμε πρώτα την προφορική τροπολογία. Κύριε Αντζελίδη, όχι δεν θέλετε το λόγο. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν ολόκληρο το ψήφισμα. Είναι ονομαστική η ψηφοφορία αυτή. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίες; Το αποτέλεσμα δείχνει ότι εγκρίνεται. Εγκρίνονται τα ψηφίσματα. And the next... And the next... Τελευταίο ε, θέμα. Επτά προτάσεις ψηφισμάτων για το Ιράν και ιδιαίτερος η υπόθεση της Νασρίν Σότουντε. Πάλι θα ψηφίσουμε στο σύνολό τους τα ψηφίσματα με ονομαστική ψηφοφορία η οποία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρας. Εγκρίνονται και πάλι με 79 ψήφους υπέρ, 0 κατά. Έχω ορισμένες ανακοινώσεις. πρόταση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά θα προσαρτηθούν στα πρακτικά της παρούσης συνεδριάσεως. Δίνεται τρίμηνη προθεσμία από αύριο